Meine sehr geehrten Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος μέχρι την ε, εκδήλωση που έχουμε σε 15 λεπτά από τώρα την παρηγενική συνεδρίαση και το υπόλοιπο θα έρθει μετά. Λοιπόν, ε, πολιτική συνοχή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην έκθεση για την έκθεση Μάριε. βελτιστοποίηση ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχων από και των περιοχών. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην έκθεση. Ορίστε. Έκθεση Τόιρερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έκθεση Ντεμπάκερ. Τον λόγο έχει ο εισηγητής. Κύριε Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ. Ε, από πλευρά τη Άλντε θέλω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για σήμερα ε, και για αυτήν την ε, σύνοδο σύμφωνα με την διάταξη 177 του καταστατικού. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος αναβολής, ποιος θα μιλήσει.